Ευχαριστούμε τη δημόσια διοίκηση. Ελπίζουμε ότι με αυτό το ψήφισμα η Ουκρανία θα βοηθηθεί για να ακολουθήσει τον οδό των οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Ευχαριστούμε. Η κυρία Πίνκε Βιτσιούτε. Ευχαριστώ πολύ